Καλημέρα σας συνάδελφοι. Ξεκινάμε με την κοινή συνεδρίαση ΕΚΟΝ ΑΦΚΟ. Είναι χαρά μου να συμπροεδρεύω με την Ντανούτα Χούμπνερ. Φαντάζομαι ότι συμφωνείτε να εγκρίνουμε τα πρακτικά, την ημερήσια διάταξη. Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις. Ωραία. Οπότε να περάσουμε απευθείας στο βασικό σημείο. Τροπολογία του άρθρου 22 για το σύστημα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ένα πολύ σημαντικό θέμα που σκοπό έχει αναλλάξει ένα άρθρο του εσωτερικού κανονισμού της Εσωτερικής Κεντρικής Τράπεζας, κάτι που σχετίζεται άμεσα και με άλλες ε, περιπτώσεις. Η Ντανούτα είναι η συνεισηγήτρια μαζί με τον κύριο Μάτο και θέλω να σου δώσω ευθύ αμέσω το λόγο Ντανούτα Ευχαριστώ, ευχαριστώ και όσου ήρθαν σήμερα το πρωί εκ μέρου της Επιτροπής άφκο. Όπως είπε μόλι ο Ρομπέρτο, σήμερα μιλάμε για το άρθρο 22 και την τροποποίησή του. Απλώς να θυμίσω σε όλους μας ότι στις 22 Ιουνίου πέρσι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εξέδωσε σύσταση για απόφαση του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το 22, άρθρο 22 του εσωτερικού της κανονισμού. Συμπλήρωμα στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 13 Ιουνίου 2017 για την τροποποίηση της, ε, του άρθρου αυτού που αφορά την εποπτεία των CCP, των κεντρικών αντισυμβαλωμένων κάτι που είναι απαραίτητο ώστε να ε, συμμετέχουν όλες οι τράπεζες. Η Κεντρική Αντισυμβαλόμενη και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ε, εντόπισαν δύο αίτια για αυτόν τον αυξημένο ρόλο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Η Κεντρική Αντισυμβαλόμενη είχαν αυξημένη εμβέλεια και διάσταση στο ρόλο τους και ευρωπαϊκός και διεθνώς, κάτι που μπορεί να προκαλέσει κινδύνους που να επηρεάσουν το όλο σύστημα και το σύστημα πληρωμών, καθώς και την εφαρμογή των νομισματικών πολιτικών. Έπειτα σημειώνεται ότι με την απομάκρυνση, την απόσταση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα υπάρξει αντίκτυπο στις επιδόσεις των συστημάτων των κρατών μελών καθώς και των κεντρικών τραπεζών ε, για την έκδοση του ευρώ. Αυτό είναι η αρχή. Η απαρχή αυτού του θέματος και βεβαίως είναι σαφές ότι αυτή τη στιγμή το σύστημα των Ευρωπαϊκών Κεντρικών Τραπεζών και της ΕΚΤ στη σημερινή του μορφή δεν θα επιτρέψει στο ευρωπαϊκό σύστημα να αναλάβει τις ευθύνες που προβλέπονται στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό συνδέεται με την απόφαση του 2015 του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου βάσει της οποίας η ΕΚΤ δεν έχει ρυθμιστικές αρμοδιότητες για αυτά τα οικονομικά εργαλεία. Γι' αυτό ξεκίνησε όλη αυτή η διαδικασία και προκειμένου να αναλάβει και να φέρει πέρα στις νέες της αρμοδιότητες η ΕΚΤ πρότεινε αυτήν την αναθεώρηση του εσωτερικού της ε, κανονισμού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε μια γνωμοδότηση σε σχέση με την αλλαγή αυτή στον εσωτερικό κανονισμό και πρότεινε ακριβώς την ε, αναθεώρηση του καταστατικού της ΕΚΤ για να αντικατοπτρίζεται στο νομικό πλαίσιο του ιστορικού κανονισμού της ΕΚΤ και αυτή η αλλαγή και εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εδώ βρισκόμαστε σήμερα. Είμαστε στην πρώτη ανταλλαγή των απόψεών μας και δύο κοινοβουλευτικές επιτροπές μελετούν αυτό το θέμα όχι μόνο από την σκοπιά της ουσίας αλλά και της θεσμικής για να μην πω συνταγματικής νομοθετικής της ε, σημασίας. Πρέπει και αυτά να ληφθούν υπόψη. Και θέλω να κάνω δύο παρατηρήσεις για αυτήν την ε, θεσμική νομοθετική προοπτική και έπειτα επί της ουσίας. Το πρώτο στοιχείο αυτής της διοργανωτικής διάστασης του θέματος έχει να κάνει με το ότι πρέπει να διαφυλάξουμε την θεσμική ισορροπία, την ισορροπία που ήδη προβλέπεται από τις συνθήκες και τον τρόπο που η Ευρωπαϊκή Ένωση λειτουργεί. Πρέπει να βεβαιωθούμε ότι οι αρμοδιότητες της ΕΚΤ να ε, λαμβάνει αποφάσεις σε έναν χώρο που τα άλλα θεσμικά όργανα, ως νομοθέτες, έχουν επίσης τη δυνατότητα να νομοθετούν. Πρέπει να διαφυλαχθεί. Πρέπει λοιπόν να ε, σεβαστούμε την αρμοδιότητα όλων των εμπλεκομένων φορέων και την παράλληλη ανάδυση συγκρούσεων κανόνων ή αντιφάσεων στους κανόνες. Πρέπει να το φροντίσουμε αυτό για να μην υπάρχουν ε, προσκόμματα στις αρμοδιότητες των θεσμικών οργάνων. Και έπειτα, ως προς την ε, διοργανωτική αυτή σκοπιά, θα πρέπει να διαφυλάξουμε το, την έκβαση των διαπραγματεύσεων για τον ιστορικό κανονισμό της ΕΚΤ και να παραμείνει συνεπής με το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων για την τροποποίηση της ε, γνωμοδότησης ιδίας πρωτοβουλίας, αυτό που τώρα τροποποιούμε. Γι' αυτό επιλέξαμε ένα σχετικό χρονοδιάγραμμα και για τα δύο θέματα, ώστε οι συζητήσεις για την ΉΜΗ να ε, συνδυαστούν με τις τροπολογίες στον ιστορικό κανονισμό και οι δύο κανόνες, ε, τα δύο σύνολα κανόνων να συμβαδίσουν, να είναι απολύτως συνεπή. Δεν σημαίνει βεβαίως ότι θα υπάρξει απόλυτη ευθυγράμμιση, διότι μιλάμε για νομικούς κανόνες και αυτή είναι η δεύτερη παρατηρήσή μου, η εράρχηση των κανόνων που πρέπει να λάβουμε υπόψη. Ο εσωτερικός κανονισμός υπερέχει υπερτερεί είναι το ανώτατο επίπεδο κανόνων νομικών ω προ τι αρμοδιότητε τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Και υπ' αυτήν την έννοια μπορεί να θεωρηθεί, να θεωρηθεί λέξη και Είναι ένα γενικός, γενικό πλαίσιο. Λέξ πεθιάλη είναι η ήμη ε, που ασχολείται με το συγκεκριμένο θέμα την εποπτεία των κεντρικών αντισυμβαλλομένων Γι' αυτό χρειάζεται και νομική βεβαιότητα ώστε πρακτικός να ελεγχθεί το πεδίο αρμοδιοτήτων της ΕΚΤ και να υπάρχει μια λογική προσέγγιση. Αλλά δεν μπορεί να γίνει στον εσωτερικό κανονισμό με έναν κατάλογο, ο οποίος, κανόνων, ο οποίος να είναι περιοριστικός, να είναι ε, ρυθμιστικός. Ο ο κανονισμός, το καταστατικό της τράπεζας δεν ε, είναι βέβαιο ότι θα αποκλείσει την αλλαγή των κανόνων στην ΙΜΗ. Ως συνήθως λοιπόν στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτήν την αντίφαση μεταξύ της ευελιξίας και της προβλεψιμότητας των κανόνων και των συζητήσεών μας. Ε, θέλουμε νομική βεβαιότητα καθορίζοντας σωστά τις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ώστε το σύστημα να μπορεί να αντιμετωπίσει και απρόσμενες εξελίξεις. ως την πρόοδο του σχεδίου έκθεσης και τις απόψεις μου επί της ουσίας, θα ήθελα να προτείνω η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η τροποποίηση όπως έχει προταθεί πέρσι, να τροποποιηθεί έτσι περαιτέρω με την δική μας παρέμβαση, ώστε οι νέες αρμοδιότητες που ανατίθενται στην ΕΚΤ να ασκούνται με τρόπο που να συνάδει με αυτά που έχουν εγκρίνει οι συνομοθέτες. Κατά δεύτερον, θα πρότενα πρακτικώς να περιοριστεί το πεδίο αρμοδιοτήτων της ΕΚΤ συμπεριλαμβάνοντας ε, ε, έναν ευρύ κατάλογο τομέων όπως η ε, ρευστότητα, οι οριμάνσεις και, άλλα τέτοια, και άλλες τέτοιες περιπτώσεις όπου να μπορεί να παρέμβει η ΕΚΤ και Επίσης κάτι που είναι εξίσου σημαντικό για την πρόοδο επί της ουσίας είναι να συμπεριλάβουμε διατάξεις για τις επίγουσες ε, ανάγκες, έκτακτες αρμοδιότητες για την Κεντρική Τράπεζα που να επιτρέπουν στην ΕΚΤ να αντιμετωπίσει καταστάσεις όπου το σύστημα των χρηματοπιστωτικών εργαλείων επιτρέπει να αντιμετωπιστούν απρόσμενοι κίνδυνοι που μπορεί να βλάψουν το χρηματοοικονομικό σύστημα. Αυτά ήθελα να πω και βεβαίως να γνωρίζετε ότι υπάρχει μια διαδικασία με κάποιες ε, ανάπαυλες βεβαίως στο Συμβούλιο που είναι σε εξέλιξη. Θα πρέπει λοιπόν να παρακολουθούμε πώς κινείται και ο συνομοθέτης. Ε, πρόεδρος, ευχαριστούμε. Ντανούτα. Και τώρα ο συνεισηγητής, κύριος Μάτο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε για αυτό το πολύ σημαντικό θέμα που μας μιλήσατε. Προσυπογράφω όλα όσα είπε η, συνεισυγήτρια η που είναι και πολύ δήμον για αυτό το θέμα. Αυτό που θα ήθελα να πω είναι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να αποκτήσει αρμοδιότητα για να απαιτήσει την λήψη διορθωτικών μέτρων σε στενή συνεργασία με τις υπόλοιπες αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην πρόταση λέμε ότι όταν είναι απαραίτητο, προκειμένου να προστατεύσουμε την σταθερότητα της Ευρωζώνης, να υπάρχουν και νομοθετικές αρμοδιότητες για να ληφθούν επιπλέον μέτρα σε σχέση με τους κεντρικούς αντισυμβαλόμενους για συναλλαγές οι οποίες γίνονται σε ευρώ. Αυτό το νέο καθήκον θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για τους σκοπούς της ενίας νομισματικής πολιτικής, για τους σκοπούς της ΟΝΕ. Για να μπορεί δηλαδή η ΕΚΤ να παίζει αυτό το ρόλο στον τομέα της ΟΝΕ. Συμφωνούμε λοιπόν με τη σύσταση της ΕΚΤΑ. Πρέπει να έχει μεγαλύτερο ρόλο στη ρύθμιση των ε, συστημάτων ε, εκαθάρισης, όμως η Κομισιόν ε, πρότεινε και κάποιες προσαρμογές σε σχέση με την πρόταση της ΕΚΤ και τα είπε όλα αυτά η Ντανούτα πολύ ξεκάθαρα για να υπάρχει συνέπεια ανάμεσα στις αρμοδιότητες της ΕΚΤ, της Κομισιόν, του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου σε ό,τι αφορά τα συστήματα εκαθάρισης. Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας το ΕΜΙΡ 2,2 Αυτή η πρόταση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σηματοδοτεί μια πολύ σημαντική αλλαγή του καταστατικού της και ελπίζουμε ότι θα μπορεί από εδώ και πέρα να εκπληρώνει πολύ καλύτερα τις α, λειτουργίες της Αυτή τη στιγμή οι κεντρικοί αντισυμβαλόμενοι ρυθμίζονται καλά χάρη στα μέτρα τα οποία έχουν ε, υιοθετηθεί μετά από την ε, χρηματοπιστωτική κρίση την κατάλληλη χρονική στιγμή. Σίγουρα όμως πρέπει να γίνουν και κάποιες επιπλέον αλλαγές για να εξασφαλίσουμε μια πιο συνεπή εποπτεία των ε, κεντρικών αντισυμβαλόμενων στην Ευρώπη και στις τρίτες χώρες. Ένα από τα τρία στοιχεία που, που είπε η Ντανούτα είναι οι δυσκολίες που προκύπτουν από κάποια κατεπήγοντα θέματα σε σχέση με τις νέες ε, αρμοδιότητες των ε, συνομοθετών σε αυτό το πιο ευρύ τομέα θεμάτων που συζητάμε σήμερα. Γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει να δοθούν μεγαλύτερες αρμοδιότητες στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για τους κεντρικούς αντισυμβαλόμενους, γιατί αυτό έχει γίνει ένα πολύ σημαντικό θέμα στις μέρες μας όλο και, θα έχει και όλο και μεγαλύτερη ε, σημασία και επιπλέον ε, μην ξεχνάμε ότι πρέπει να δούμε και το θέμα του Ηνωμένου Βασιλείου το οποίο θα φύγει ως ο Νούμπο ε, και τη θέση που θα έχει σε όλο αυτό το σύστημα. Όπως είπε πολύ σωστά η ένα βασικό θέμα είναι η συνταγματική αναπροσαρμογή Περιμένουμε λοιπόν τη γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας για να μας μιλήσουν για τα συνταγματικά θέματα. Ευχαριστώ. Ο σκιώδης εισηγητές της, της ΕΚΟΝ, η κυρία Περβάνς Μπερές. Είμαι η σκιώδης εισηγήτρια και στις δύο επιτροπές. Άρα θα κερδίσουμε λίγο χρόνο αφού είμαι και στις δύο επιτροπές. Σας ευχαριστώ για το ραντεβού που μας δώσατε για ένα θέμα το οποίο το περιμέναμε. Ε, έπρεπε να γίνει δεδομένου του ΕΜΗΡ 2,2. Ε, Υπάρχουν διάφορα θέματα τα οποία ζητήσαμε να μας ξεκαθαρίσει η νομική μας υπηρεσία. Αυτά τα θέματα Του θα ρωτήσαμε πριν από δύο μήνες, ε, αν δεν απατώμε, και δεν μας έχουν απαντήσει καθόλου, ούτε κατά διάνοια. Τα νομικά θέματα που ζητάμε να διευκρινιστούν είναι για πολύ σημαντικά θέματα. Η νομική υπηρεσία όλων των άλλων θεσμικών οργάνων έχουν ανασκουμποθεί. Δεν θέλω να προκαλέσω τον ανταγωνισμό μεταξύ νομικών υπηρεσιών, αλλά σε τέτοιε καταστάσει ποια είναι η πρακτική. Μπορεί να είναι ενδιαφέρον, εν πάση όχι να κάνουμε τώρα μια, έναν ανταγωνισμό και μια άμυλα, ας πούμε, αλλά μια συμπληρωματικότητα να υπάρχει ε, από τις, ε, χάρη στις συνεισφορές των νομικών υπηρεσιών. Ελπίζω να υποφεληθούμε από αυτή τη νομική συμβουλή εγκαίρως. Επί της ουσίας τώρα. Καθορίζεται από τρεις άξονες καταρχάς την απόφαση του δικαστηρίου η οποία αφορά την ε, ΕΚΤ και υποχρεώνει την ΕΚΤ καθώς και το νομοθέτη να προβεί στο, στην αλλαγή του καταστατικού ε, λαμβάνοντας υπόψη και τα δύο επόμενα στοιχεία που θα αναφέρω. Καταρχάς ότι είναι όλο και πιο σημαντική η κεντρική αντισυμβαλόμενη και έχουν συστημική σημασία λόγω της ε, μεταβίβασης της ε, λήψης ε, κινδύνου μετά από τις εξελίξεις της αγοράς και το πώς αντιμετώπισε η αγορά την κρίση και τρίτον της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από, από την Ευρωπαϊκή Ένωση που θε, ένα θέμα εποπτείας και τρόπου λειτουργίας των κεντρικών αντισυμβαλόμενων που βρίσκονται εκτός της ε, αρμοδιότητας ή της δικαιοδοσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα, επί της ουσίας της υπόθεσης, νομίζω ότι το δικό μας όργανο πάντα μίλησε για την εξαρτησία της ΕΚΤ και κανένας στη Γαλλία τουλάχιστον δεν αμφισβητεί αυτή την ανεξαρτησία, μια και η εντολή της ΕΚΤ ήταν πάντα σαφής. Το θέμα όμως του πώς θα ερμηνεύσουμε μία δραστηριότητα της ΕΚΤ, η οποία μπορεί να εξελίσσεται λόγω της εξέλιξης της νομοθεσίας, ε, θέτει ένα πρόβλημα θεμητό νομίζω. Και έχει δίκιο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα που ανησυχεί για αυτή την πτυχή. Την τροποποίηση του άρθρου 22, δηλαδή όπως το προτείνει η Κομισιόν. Από αυτά που λέει η Ντανούτα καταλαβαίνω ότι μία λύση που προτάθηκε μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα. Δηλαδή να βάλουμε στο άρθρο 22 ε, μία αντιγραφή αυτού που υπάρχει στο ΕΜΥΡ 2. Ποιοι είναι δηλαδή οι συγκεκριμένοι τομεί επί των οποίων χρειαζόμαστε ε, την άμεση παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, αντιγράφοντάς το από το ΕΜΥΡ 2.2 από το ΕΜΙΡ 2 μάλλον, για να εξασφαλίσουμε τη σταθερότητα του συστήματος πληρωμών, γιατί αυτό είναι το βασικό θέμα. Και είναι και η βασική αρμοδιότητα της ΕΚΤ. Εγώ είμαι ανοιχτή να έχουμε μια διατύπωση που να βασίζεται σε κάποιες αρχές, αλλά νομίζω ότι αυτό είναι το σημείο ισορροπίας. Νομίζω ότι θα πρέπει να συμφωνήσουμε επί της αρχής, δηλαδή ότι χρειαζόμαστε να προχωρήσουμε παράλληλα με το ΕΜΙΡ 2, δηλαδή άρθρο 22 και ΕΜΙΡ 2 και τα δύο μαζί. 2. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν μπορεί να αφήνει την, ε, το καταστατικό της να καθορίζεται από ε, μια νομοθεσία επίπεδου 2 που θα την ε, διαμόρφωνε από μέρα σε μέρα και τρίτον χρειαζόμαστε μια ξεκάθαρη εικόνα για τη λειτουργία και τα πρότυπα των ρυθμίσεων και των κανόνων επί των οποίων και βάσει των οποίων παρεμβαίνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Να προσθέσω και ένα τέταρτο. Ο τρόπος με τον οποίο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ασχολήθηκε με αυτή την πρόταση κανονισμού. Πώς παρεμβαίνει. Βλέπω τον πρόεδρο που με κοιτάζει. Εσείς και εγώ και εμείς ε, θυμόμαστε πώς εξελίχθηκαν οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σε αυτό το τομέα, όπου τότε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε ζητήσει να μπορεί να παρεμβαίνει. Θα πρέπει λοιπόν να κοιτάξουμε και αυτή την πτυχή στην πρόταση. Γιατί μέχρι στιγμής δεν άκουσα τους ε, δύο εισηγητές να το αναφέρουν, αλλά είμαι σίγουρη ότι το έχουν στο μυαλό τους. Um, Ευχαριστούμε. Από το ECR. Εκπροσωπεί τον κύριο Λούνς. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Οπωσδήποτε δεν εκφράζω τις δικές μου απόψεις αλλά του κυρίου Λούντς, ο οποίος ε, κολλείεται. Μου έχει γράψει όμως κάποιες σημειώσεις, τις οποίες θα διαβάσω. εξήγησαν οι προηγούμενοι μιλητές στο πλαίσιο της έκθεσης, δεν θα τα επαναλάβω. Αλλά ο Σάντερ Λούντς αντιλαμβάνεται ότι υπάρχει κάποια νομική ανάγκη να τροποποιηθεί το άρθρο 22 των ε, καταστατικών ε, της ΕΚΤ για να μπορέσει να ρυθμιστεί η πολιτική του CCP και θεωρεί ότι θα πρέπει μια πολιτική αυτή να ασκείται στο πλαίσιο της πολιτικής της ΕΚΤ και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Αυτά που ξέρουμε συνδέονται με την αναθεώρηση του ΕΜΗΡ και ο κύριος Λιόνς λέει ότι θα πρέπει να περιοριστούμε σε αυτό. Θα ήθελα να τονίσει ότι οι αλλαγές στο άρθρο 22 χρειάζονται για να υπάρχουν τα απαραίτητα νομικά εργαλεία έτσι ώστε να εκπληρωθούν τα όσα αναφέρονται στον ΕΜΗΡ και άλλους κανονισμούς. Και καλωσορίζεται ότι υπάρχει γνωμοδότηση από την νομική υπηρεσία την οποία αναμένουμε και αναμένει την ερμηνεία που θα δώσει η νομική υπηρεσία. Και αναμένει βεβαίως το σχέδιο έκθεσης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ από την ΑΦΚΟ και το Ισιάρο, Ο κύριος με Σμίτ απουσιάζει. Α, εδώ είστε. Μάλιστα, μα δεν θέλετε να μιλήσετε όμως. Οπότε μπορούμε να περάσουμε στην ΑΦΚΟ. Ο κύριος Γκέρνσεν εδώ. Ή δεν βλέπω καλά. Κύριε Γέτζακ, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Υπάρχει η απόφαση του δικαστηρίου για το άρθρο 22 του καταστατικού της εκτε και δεδομένου του ρόλου που παίζει στο περιβάλλον ε, το τωρινό και την πιθανή συστημική φύση κάποιων κεντρικών αντισυμβαλωμένων θα πρέπει η να μπορεί να έκπληρουν τα καθήκοντά τη για να διασφαλίσει την νομισματική σταθερότητα. Οπότε, σε γενικέ γραμμέ, η ομάδα μα στηρίζει το αίτημα της ΕΚΤ για την αλλαγή στο άρθρο 22. Παρ' όλα αυτά, όπως είπε και η Κομισιόν, η αναθεώρηση του άρθρου 22 σημαίνει ότι υπάρχει κίνδυνος να επεκταθεί υπερβολικά το πεδίο εφαρμογής ε, και να έρθει έτσι η ΕΚΤ σε σύγκριση με κανονισμούς που έχει εγκρίνει το Συμβούλιο ή το Κοινοβουλίο. Πρέπει να αποφευχθεί αυτή η κατάσταση και θα πρέπει ακριβώς να ορίσουμε όσο πιο στενά γίνεται το πεδίο εφαρμογή για να μπορεί η να κάνει καλύτερα την δουλειά της χωρίς να εμπλέκεται σε τομείς αρμοδιότητας των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σβέν ναι, Σας ευχαριστώ. Σε γενικές γραμμές στηρίζουμε την ε, σύσταση της ΕΚΤ και θεωρούμε ότι είχαν υπάρξει κάποιες χρήσιμες ε, ευκρινήσεις που είχαν γίνει από την Κομισιόν. Δεδομένων δε των ε, πρόσφατων αποφάσεων του δικαστηρίου όλα αυτά είναι λογικά και προφανώς συμφωνούμε με την άποψη της Κομισιόν να επιμείνουμε ότι αυτά πρέπει να συμμορφώνονται και με το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο. Για τις παρατηρήσεις που έκανε τώρα η συγγετριά μας και πρόεδρος της ΑΦΚΟ, η Ντανούτα, βεβαίως ε, μπορούμε να μπούμε σε περισσότερες λεπτομέρειες, αλλά θα πρέπει να επιμείνουμε ότι ο κατάλογος αυτός ε, να μην είναι κλειστός και οριστικός. Και όσον αφορά τις έκτακτες αρμοδιότητες υπάρχουν παρόμοιες τροπολογίες στο πλαίσιο του δεύτερου εμμύρ Οπότε δεν ξέρω, κάνουμε τα ίδια πράγματα δύο φορές. Ίσως θα μπορούσαμε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί κάνοντας ε, κάτι τέτοιο στην αναθεώρηση του δεύτερου εμμύρη, αλλά δεν είναι και τόσο θρησκευτικό το ζήτημα. Σε γενικές γραμμές στηρίζουμε την ε, γραμμή της ηγητρίας. Σας ευχαριστώ κύριε. Ο κύριος Βιάγκας από την ΚΟΕ. Ναι, παρακαλώ. Eh, Δεν ενημερώθηκα από την σκιώδη συγκητή μας, βρίσκεται στην Άγκρη. Απλώς, προφανώς μια ανησυχία έχουμε, δηλαδή θα πρέπει να κοιτάξουμε ότι θα συμβαδίσει η αλλαγή αυτή με την εξέλιξη του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Και πρέπει να πω και το εξής. Διαρκώς αντιμετωπίζουμε την ε, ατέρμονη δημιουργικότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος που διαρκώς μεταλλάσσεται, διαρκώς παρακάμπτει, διαρκώς ε, χρησιμοποιεί τα θεσμικά όργανα με την πρόκληση να βρίσκει νέους τρόπους να ε, προσαρμόζεται. Πρόκειται για ένα τέρας το οποίο δεν μπορούμε να ελέγξουμε και αυτή τη στιγμή έχουμε μία ακόμη μεταμορφωσή του με επιπλέον μια απόφαση του δικαστηρίου Έχουμε λοιπόν προφανώς επιφύλαξη, διότι στο μέλλον το θέμα αυτό θα πρέπει να τεθεί σωστά. Η αύξηση του ε, παράλληλου τραπεζικού τομέα, το χρηματοπιστωτικό σύστημα με τα πλοκάμια του θα πρέπει λοιπόν να κοιτάξουμε με σύνεση το όλο θέμα και εκφράζουμε σκεπτικισμό και επιφύλαξη για την δυνατότητα να ε, διευθετήσουμε το χρηματοπιστωτικό σύστημα χωρίς να κοιτάζουμε τα γενεσιουργά αίτια των προβλημάτων και διαρκώς να αναζητούμε ε, πιο προηγμένους τρόπους και πιο ε, εξελιγμένους για να ελέγξουμε τον εξέλιγκτον. Δεν βλέπω συναδέλφους από την EFTD, δεν βλέπω τον κύριο Καστάλντο. Κύριε Μονό, Ο κύριος Μαν. <clears throat> Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι για το ότι υπάρχει μεγάλη συνένεση να πούμε ότι πρέπει να υπάρξει μια αλλαγή του καθεστώτος ε, σύμφωνα με την απόφαση του 10 για το άρθρο 22. Και χαίρομαι για αυτά τα οποία είπαν οι προλελήσαντες. Τώρα για το αν είναι σημαντική η αλλαγή ε, πρέπει να είμαστε νομίζω πολύ σαφείς ε, στην παραγραφό 22. Η ερώτησή μου στην ε, Ντανούτα είναι η εξής. εντάξει, μπορεί να μην υπάρχει καμία αφιβολία για την εξαρτησία της ΕΚΤ, αλλά όταν θα έχει τις νέες αρμοδιότητες, πώς μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι θα χρησιμοποιηθούν μόνο για νομισματικούς σκοπούς να επικεντρωθεί δηλαδή μόνο σε αυτό το θέμα. Αυτό με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Κατά εξαίρεση, επειδή είστε δυσκείοδες και στα δύο Ναι, ναι, επειδή κάτι ξέχασα. Δεν ξέρω αν είναι εδώ πέρα κάποιος από το Συμβούλιο ή μπορεί να μας πει η Κομισιόν κάτι για το τι άποψη έχει το Συμβούλιο. για να έχουμε μια εικόνα του τι συμβαίνει. Δεν υπάρχει κανείς. Ε, νομίζω μπορούμε να ακούσουμε την Κομισιόν. Εξ όσων γνωρίζω δεν συμβαίνει τίποτα στο Συμβούλιο, αλλά ίσως η Κομισιόν να έχει νεότερα στοιχεία. Δεν ξέρω ποιος είναι εκεί. Ποιος είστε? Ο κύριος Πίεσον. Θέλετε να πείτε κάτι? Ναι, θα είμαι σύντομος, κύριε Πρόεδρε. Ναι, αλλά και για το Συμβούλιο. Ναι, ναι, απαντήστε και στην ερώτηση της κυρίας Μπερές. Πρόεδρε, θα είμαι πολύ σύντομο. Καλωσορίζουμε την πρωτοβουλία τη για τρει λόγου. Η κεντρική αντισυμβαλόμενη συστημικώ έχουν ένα και μεγαλύτερη σημασία λόγω των κινδύνων. Δεύτερο λόγο, το Brexit, που θα κάνει τι δυσκολίε μεγαλύτερε. Είναι σαφέ. Γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε αυτή την τροποποίηση για να έχουν οι κεντρικέ τράπεζε ενισχυμένο ρόλο. Επίσης, ο τρίτος λόγος είναι ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο είναι πολύ σαφέ. Έχει αρμοδιότητε η ΕΚΤ στο πεδίο του συστήματο πληρωμών, αλλά όχι σε όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία. Εάν θέλουμε να εγκριθεί το ΕΜΗΡ, εάν θέλουμε να έχει αυτέ τι νέε αρμοδιότητες η ΕΚΤ, για να μπορεί να τι ασκήσει. Θα πρέπει να ε, τροποποιηθεί το άρθρο 22 του καταστατικού. Είναι πολύ σαφέ. Όμω επίση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει καταστήσει σαφέ ότι πρέπει να είμαστε συνεπεί και να πλαισιώσουμε τι ρυθμιστικέ αρμοδιότητε τη ΕΚΤ για να μην υπάρξει σύγκρουση και αντιφάσει στου κανόνε που προκύπτουν από αυτό το σώμα και από το Συμβούλιο. Θα πρέπει να έχουμε υπόψη ότι το καταστατικό τη ΕΚΤ στι αλλαγέ του πρέπει να έχει την σωστή εξισορρόπηση δεν υπάρχει άλλο είδου ιεραρχία και δεν επηρεάζεται και η ανεξαρτησία της ΕΚΤ. Θα πρέπει η διατύπωσή μας να τα σεβαστεί όλα αυτά. Η σχετική δουλειά στο Συμβούλιο συνεχίζεται σε 18 λεπτά. Το ρολόι προχωρά. Σε 18 λεπτά θα ξανασυναντηθεί το Συμβούλιο, η ομάδα εργασία και σε γενικές γραμμέ υπάρχει συμφωνία ότι το, το θέμα τη ΕΚΤ για τις νέες της αρμοδιότητες είναι λογικό. Το Συμβούλιο συζητά συγκεκριμένου τομεί όπου μπορεί αυτέ οι αρμοδιότητε να ασκούνται, όμω δεν υπάρχει στο Συμβούλιο διαφωνία μεταξύ των κρατών μελών ότι το θέμα τη ΕΚΤ θα πρέπει να ε, δημιουργήσει πρόβλημα. Okay, so... Ευχαριστούμε. Είσαι γήτρια. Πολύ σύντομα. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει ευρεία πλειοψηφία για να προχωρήσουμε με την τροποποίηση του άρθρου 22. Υπάρχει στήριξη. Φαίνεται όλα τα θεσμικά όργανα να κινούμαστε στην ίδια κατεύθυνση. Κατά δεύτερον, νομίζω ότι υπάρχει αρκετή εμπιστοποίηση στο Κοινοβούλιο για να βλέπουμε ότι η θεσμική ισορροπία, που εν μέρει αναφέρθηκε και πάλι, ο ρόλο των θεσμικών οργάνων, ιδίω των συνομοθετών, δεν πρέπει εδώ να ε, διαταραχθεί. Καταλαβαίνουμε αυτή την πρόκληση και μετά χρειάζεται και η σωστή διατύπωση. Πρέπει να σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μην ανοίγει την πόρτα σε τίποτε το ανεπιθύμητο. να μην επηρεαστεί ο ρόλο ενό τόσο και σημαντικού θεσμικού οργάνου τη ΕΚΤ, να μπορεί και στο μέλλον να ενεργεί αποτελεσματικά συγκεκριμένου τομεί. Πρέπει εδώ να έχουμε υπόψη μας και το μέλλον ότι υπάρχουν καταστάσεις που μπορεί να προκύψουν και που σήμερα δεν τις γνωρίζουμε. Η αλλαγή στο καταστατικό λοιπόν δεν είναι και κάτι που μπορεί να γίνεται όποτε μας έρχεται. Γι' αυτό θα πρέπει να βρούμε μια ισορροπία μεταξύ των επιπλέον αρμοδιοτήτων που μπορεί να αντιμετωπίσουν οι συνομοθέτες. Ευχαριστώ πολύ λοιπόν Πρόεδρε της ΕΚΟΝ, ευχαριστούμε πολύ για τη δυνατότητα που μας δώσατε. Να δώσω το λόγο και στον άλλο συνεισηγητή, τον κύριο Μάτο. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους για τις παρεμβάσεις σας. Ε, προκύπτει ξεκάθαρα η ανάγκη για αυτή τη μεταρρύθμιση, την οποία, στην οποία θα εμπλακούμε όλοι. Περιμένουμε αυτή την, την ε, νομική γνωμοδότηση που μας χρειάζεται και όπως είπα και στην πρώτη μου παρέμβαση, είναι πολύ σημαντικά δύο πράγματα. Η σημασία των κεντρικών αντισυμβαλλόμενων και το Brexit. Είμαι πεπισμένος ότι όλοι μαζί από κοινού θα καταφέρουμε να φτιάξουμε μια καλή έκθεση. Το χρονοδιάγραμμα. Να σας πω ποιο είναι. Μισό λεπτό. Πρέπει να επιβεβαιωθεί ένα βασικό θέμα. Καταρχάς θέλουμε τη νομική γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας. Την παρακινούμε να ολοκληρώσει την γνωμοδότησή της, γιατί όλοι έχουμε εντοπίσει τα προβλήματα, αλλά όχι τις, λύση, τις λύσεις. Έχουμε ακόμα χρόνο για να μας δώσει κάτι η νομική υπηρεσία. Το χρειαζόμαστε αυτό το κάτι. Προς το παρόν, λοιπόν, στις 28 Μαρτίου θα ετοιμάσουμε την ε, γνωμοδότηση. 24 ε, Απριλίου θα την παρουσιάσουμε. 2 ε, Μαΐου τις τροπολογίες. Θα εξετάσουμε τροπολογίες 24 Μαΐου και στη, θα ψηφίσουμε στις 19 Ιουνίου. Άρα για την ε, προθεσμία ε, της έκθεσης, μέχρι την, από την ετοιμασία μέχρι την παρουσίαση, καλό είναι να έχουμε και λίγο χρόνο. Δεν θέλουμε να αλλάξουμε την ημερομηνία ε, για την ετοιμασία της ε, γνωμοδότησης, ε, αλλά γι' αυτό χρειαζόμαστε την νομική γνωμοδότηση. Πολύ ωραία. Τελειώσαμε αυτή την σύντομη σύνοδο, αλλά πολύ επωφελή και πάμε σε σύνθεση έκον.